Buongiorno. Καλημέρα. Cominciamo con eh, le informazioni sulla riunione dei coordinatori. Να αρχίσουμε πληροφορώντας σας σχετικά με τη συνεδρίαση των συντονιστών εχθές. <coughs> Αποφασίσαμε σε ένα σωρό σημεία για την απαλλαγή της Κομισιόν για το 2008 με εισηγητή τον κύριο Λιμπεράσκη. Όσον αφορά στην απαλλαγή του 2009 ο κύριος Χατζημαρκάκης ε, είναι ο εισηγητής σχετικά με την απαλλαγή για το 2009 του Κοινοβουλίου είναι ο κύριος Ήταλα για την απαλλαγή του 2009 για τα άλλα όργανα, ο κύριος Ριβελίν είναι ο εισηγητής. Για την απαλλαγή 2009 οργανισμοί, ο κύριος Σταυρακάκης. Σχετικά με τον Ιρλανδό υποψήφιο για το ελεγκτικό συνέδριο είναι η κυρία Γιάλα Σέντερ. Πρόταση κανονισμού τροποποίησης του Συμβουλίου για τον δημοσιονομικό κανονισμό για τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης ο κύριος Ριβελίνη που ορίστηκε εισηγητής και ο πρόεδρος μαζί με τον πρόεδρο της Επιτροπής Προϋπολογισμού θα στείλει μία επιστολή για το άρθρο 50 σχετικά με τις αρμοδιότητες των δύο επιτροπών. Για τη γνωμοδότηση της Επιτροπής μας στην ΑΦΚΟ για τη διαθεσμική συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Συμβουλίου και Κομισιών για τη συνεργασία για τα δημοσιονομικά θα τα αναλάβει ο πρόεδρος, δηλαδή εγώ. Ο κύριος Κάλφιν ορίστηκε της, ε, εισηγητής της ΚΟΝΤ για την απόφαση του Συμβουλίου για την οργάνωση των εξωτερικών υπηρεσιών και ως εκπρόσωπος της ε, Επιτροπής της ε, Κοκομπού για την μεικτή ομάδα εργασίας. Τώρα για τις άλλες πλευρές της των εξωτερικών υπηρεσιών, ο για τον δημοσιονομικό κανονισμό ο κύριος Ριβελίνη ανέλαβε και όσον αφορά για το καταστατικό των υπαλλήλων η κυρία Χέρτσοκ και ο κύριος Μπάλτσεβιτς για τον διορθωτικό προπολογισμό. Τώρα για την απαλλαγή το 2009 για την Κομισιόν, ο κύριος Χατζημαρκάκης, για το Κοινοβούλιο ο κύριος Ήταλα, ο κύριος Ριβελίνη για, τα υπόλοιπη, για τους υπόλοιπους οργανισμούς και ο κύριος Σταυρακάκης για τους άλλους οργανισμούς. Τώρα, για τον διορισμό του Διευθυντή της Όλαφ, το αναπληρωτή διευθυντή της Όλαφ, αποφάσισαν οι συντονιστές ότι δεν χρειάζεται να γίνει συζήτηση με τον κύριο Ήλετ, όπως είχαν ζητήσει δηλαδή στη διάσκεψη των πολιτικών ομάδων. ορίστηκε το, το τελικό πρόγραμμα για την επίσκεψη στην Ελλάδα από τις 27 ως τις 29 Απριλίου. Θα συμμετέχει και ο κύριος Χατζη Μαρκάκης Ιδίες Δαπάνες, όπως και ο κύριος Ντελάνγκε ο οποίος ζήτησε να συνοδεύεται από τον βοηθό του. Επίσης, ο κύριος Γκράσλε ζήτησε, ότι θα, είπε μάλλον ότι θα συμμετέχει και ο κύριος Ντεβίνο, ο, αναπληρωτ, ο αναπληρωτής διευθυντής Γεωργίας, ο υποδιευθυντής μάλλον της Γεωργίας, όπως είχε γίνει και το 2007, για την αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού θα γίνει μια κοινή ακρόαση την 1η Ιουνίου το πρωί μεταξύ της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και της Επιτροπής Προϋπολογισμών. Εγκρίθηκαν λοιπόν οι προτάσεις. Αυτά μάλλον εγκρίθηκαν. Ο κύριος Ριβελίνη θα προτείνει τους ομιλητές και ορίστηκαν επίσης και πέντε μελέτες οι οποίες μερικές συμπτύχθηκαν και οι οποίες θα υλοποιηθούν το 2010 και άλλες το 2011. Η Γραμματεία έχει μοιράσει σε όλα τα μέλη της Επιτροπής τον έλεγχο των μελετών για το 2010 οι άλλες αναβάλλονται για το 2011. Τώρα, για την αντιπροσωπεία στην Κροατία θα γίνει η επίσκεψη από τις 23 με τις 25 Ιουνίου με κοινή αντιπροσωπεία μεταξύ της ε, Κόκομπου και της Επιτροπής Προϋπολογισμών. Σχετικά με τον διάλογο για τις ε, επιτροπές ε, και των επιτρόπων εμείς ε, λάβαμε υπόψη μας την πρόταση του κυρίου Λένε εκ μέρους της διάσκεψης των Προέδρων και συμφωνήσαμε ότι θα αναβάλουμε την ακρόαση του κυρίου Σεμέτα διότι ήταν πολύ νωρίς να γίνει η ακρόαση αυτή τον Απρίλιο όπως έλεγε ο κύριος Λένε. Επίσης εμείς έχουμε φτιάξει και ένα σχεδιάγραμμα για την παρακολούθηση των δεδομένων που θα μας έρχονται από το West Wolf. Επίσης, για... Επίσης μοιράστηκε χθε στους συντονιστές ένα σημείο μας σχετικά με το διορισμό του κυρίου Φαζάκα στον... στο ελεγκτικό συνέδριο. Αυτά για τα χθεσινά στους συντονιστές. Λοιπόν, πάμε τώρα στην ε, απαλλαγή 2008, Γενικό Προπολογισμό Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Λοιπόν, πριν ψηφίσουμε, δίνω το λόγο στον Αντιπρόεδρο Στάις που είναι εισηγητή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Έχετε τον κατάλογο για την ψηφοφορία. Κάναμε τις συζητήσεις ε, και ακούσατε όλοι τα σχόλια μου όταν παρουσίασα το σχέδιο. Ε, υπήρξε θετική αντίδραση από πλευράς των συναδέλφων. Έχουμε 102 τροπολογίες. Ε, ευνηδιάστηκα από αυτό το μεγάλο αριθμό τροπολογιών, πρέπει να πω. Αλλά έχουμε δύο ακραίες θέσεις και δεν έχουμε καταφέρει ουσιαστικά να βρούμε μέση οδό. Κάποιοι θεώρησαν ότι ήμουν υπερβολικός στη διατύπωσή μου και έχουν υποβάλει διάφορες τροπολογίες για απαλληφή επιμέρους σημείων ε, της έκθεσης. Υπήρξαν βέβαια και πολλοί επικοδομητικές τροπολογίες, προσπάθησα να τις συμπεριλάβω ε, και μιλώ για τροπολογίες που έρχονται από όλες τις πολιτικές ομάδες, σοσιαλιστές, ε, γκουε, το ΕΛΚ, όλοι υπέβαλαν τροπολογίες. Ε, και σας είπα ότι υπήρχαν και διάφορες τροπολογίες ε, που προτείνουν απαλληφή σημείων. Ε, εγώ προτείνω να τις καταψηφίσετε, αν τελικά εγκριθούν. Θεωρώ ότι η έκθεση έχει σκοπό να δώσει στο management εδώ, στη διακυβέρνηση του Κοινοβουλίου, ένα καλό τρόπο να, διαχειριστούμε τα χρήματα. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να συνεχιστούν αυτές οι προσπάθειες. Δεν νομίζω ότι είναι δύσκολη η ψηφοφορία. κυρία Χέρτσοκ χθες ε, απέσυρε μια σειρά τροπολογιών. Θα ήθελα να συμφωνήσω με κάποιες από τις τροπολογίες αυτές και χτες επίσης με το ΕΛΚ και με τους σοσιαλδημοκράτες συμφωνήθηκε κυρίως σε ό,τι αφορά την παράγραφο 106 να εξευρεθεί μια αποδεκτή διατύπωση. Να προτείνω να πάρω το λόγο για να δούμε τελικά επί ποιο κειμένο θα ψηφίσουμε. Πρόεδρε, προτείνω να παρέσουμε στην ψηφοφορία. Onorevole Staes, anche per il lavoro molto impegnativo che ha svolto, quindi Ευχαριστούμε τον κύριο Στάις για τη δουλειά του. Λοιπόν, θα πάμε τώρα στην ε, ψηφοφορία, η οποία θα είναι ιδιαίτερα επίπονη. Έχετε όλοι σας, ελπίζω, την κάρτα ψηφοφορία σχετικά με την απαλλαγή για το 2008. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. approvato 21 voti favorevoli e 4 contrari. Passiamo adesso alle risoluzioni per quanto riguarda votazione. E Πάμε τώρα στα ψηφι... στο ψήφισμα. Τροπολογία, εναρχής ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Δύο. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τρία. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 18-9. Τέσσερα. Αρχίζει ψηφοφορία. Α, καταπίπτει. Συγγνώμη. Λοιπόν, πέντε. Ψηφίζουμε. Ένα λεπτό, ένα λεπτό, λέει ο πρόεδρος. Πέντε, πέντε έλεγα. Αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 25 υπέρ. Έξι. Αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 24-3. 7. αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 8. αρχιζει ψηφοφορια ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 19-8 το σκορ. 9. Έτσι όπως ορίζεται αρχίζει ψηφοφορία, πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 10 αποσύρθηκε, 11 ψηφίζουμε. Πέρας. εγκρίνεται με 27 ψήφους υπέρ, 12 αρχίζει ψηφοφορια ψηφοφορία, πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 19-8, 13 αρχίζει ψηφοφορία, πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 14. Αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας, Εγκρίνεται. 15, 16, 17 τα ψηφίζουμε αν συμφωνείτε. Αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας, Εγκρίνονται. 15, 18. Ψηφίζουμε πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 19. Ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται 22-6. 20 αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 21 αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 22 αρχίζει ψηφοφορία Πέρας ψηφοφορία. Α, καταπίπτει. 22. Η 23 αποσύρθηκε. Λοιπόν πάμε στην 24. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 25 ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 26. Ε, πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 26. Η 27. 27. Αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Η 29. Αρχίζει ψηφοφορία. Α, όχι η 29. Α, η 30, η 30. Ψηφίζουμε λοιπόν. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. 31. Αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Καταπίπτει 32. 33 αποσύρθηκε, 34 αρχής ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. 35 αποσύρθηκε, 36 αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 37 αποσύρθηκε, 38 με χωριστή ψηφοφορία. Το πρώτο του κομμάτι αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Το δεύτερο κομμάτι της 38 αρχίζει ψηφοφορία, πέρας ψηφοφορίας, απορρίφθηκε. 39 αποσύρθηκε, 40 αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 41 αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 42 αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Η γραμματεία μου λέει ότι οι σοσιαλιστές είναι παραπανήσιοι. Έχει πολλούς που ψηφίζουν για τη σοσιαλιστική ομάδα. Κάποιος από εσά πρέπει να πάει για καφέ, λέει η γραμματεία. Ναι, εντάξει πρόεδρε. Λοιπόν, για διαπιστώστε εκεί ποιος ψηφίζει στη σοσιαλιστική ομάδα Παραπανήσιος. Ο συνάδελφος Μπέρμαν ψηφίζει και θα πρέπει να φύγει η συνάδελφος Αγιάλα λόγω ανελειμμένων υποχρεώσεων. Θα είμαστε και πάλι οκτώ. Φαντάζομαι ότι είναι οκ 43, 43. Ωραία, λοιπόν, πού φτάσαμε, λέει ο πρόεδρος, 43. Ωραία. Λοιπόν, 43 ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 44. Αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. 45 ψηφίζουμε. Εγκρίνεται. 46 αρχίζει η ψηφοφορία πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται 47 αρχίζει η ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται Για να το επαληθεύσουμε γιατί το κομπιούτερ πάλι έναν παραπανίσιο. Μπα και άφησε την κάρτα στο μηχάνημα η κυρία Γιάλα. Okay. Ωραία. Ας προχωρήσουμε. Καμιά φορά τα κομπιούτερ είναι χειρότερα και από τους ανθρώπους. Πάμε λοιπόν στη 48 ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 40... Ε, α, μπερδεύτηκε ο πρόεδρος. Λοιπόν, 51. Πρώτο τμήμα, αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Α, η 51 έχει καταπέσει, λοιπόν ζητώ συγγνώμη, 52 ψηφίζουμε. Αρχίζει η ψηφοφορία, πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 53.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 Ψηφίζουμε μαζί από την 56 μέχρι και την 59 και αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 60. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτω. 61. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 62 αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 63 αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται.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 Ε, συγγνώμη, Πρόεδρε, κάτι ήθελα να ελέγξω για την 63 της κυρίας Γκρέσλερ. Δεν ήταν διαγεγραμμένη πλήρως αυτή η τροπολογία. Και κοιτώντας ε, την ε, τροπολογία της κυρίας Χέρτσοκ, αν την αν συμφωνήσω με αυτή, μπορούμε να ψηφίσουμε. Κύριε Χέρτσοκ, την αποσύρατε εσείς την ψηφοφορία, την ε, τροπολογία, συγγνώμη, αλλά εγώ θα την ε, ξαναυποβάλλω και νομίζω ότι μπορούμε να την ψηφίσουμε στην περίπτωση αυτή. Α, δηλαδή σαν να είναι προφορική η τροπολογία του κυρίου Στάς, μάλιστα. Ο κύριος να το σκεφτούμε λίγο αυτό. γιατί από όσο κατάλαβα, η τροπολογία της κυρίας Γκρέσλε αναφέρεται στο παλιό κείμενο του κυρίου Στάς, στην παράγραφο 9.29. Και η παράγραφος, η τροπολογία 64 της κυρίας ε, ε, Γκρέσλε είναι συμπλήρωμα, δηλαδή αν δεν υπάρχει κάποια αντίφαση προς το κείμενο, πρόκειται για προσθήκη, καθαρά προσθήκη αν το κάνουμε έτσι, δεν θα ισχύει ο κατάλογο ψηφοφορία, γιατί θα πρέπει πρώτα να ψηφίσουμε την πρόταση διαγραφή. Γι' αυτό λοιπόν ουσιαστικά θα δημιουργηθεί πρόβλημα στον κατάλογο ψηφοφορία, καταλαβαίνετε. Ο κύριος ε, Στάς, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να περιπλέκουμε τα πράγματα. Να προχωρήσουμε την ψηφοφορία και πάντα υπάρχει και η ολομέλεια για να υποβάλουμε ενδεχομένω άλλες τροπολογίες. Άρα μπορούμε να προχωρήσουμε με την επόμενη παράγραφο. Ωραία. 65. Αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 67. Αρχίζει ψηφοφορία. εγκρίνεται. Εβδομήντα αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. ένα αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 73 αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 74 αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 75 αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 78. Αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 80. Αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. 81 αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. 83 αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. 84 αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. 86 αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 88 αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. 89. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 91 χωριστή ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 91, αρχίζει ψηφοφορία, πέρας της ψηφοφορίας, απορρίπτεται. 92 χωριστή ψηφοφορία, πρώτο τμήμα. Α, έχει καταπέσει το πρώτο τμήμα. Δεύτερο τμήμα λοιπόν. Ωραία, ψηφίζουμε το δεύτερο τμήμα της 92, αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 93. Αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 95. Αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία εγκρίνεται. Ενενήντα Χωριστή ψηφοφορία. Το πρώτο τμήμα. Αρχής ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Αρχίζει ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας, απορρίπτεται. Τρίτο τμήμα. Αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τέταρτο τμήμα. Αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τελευταίο κομμάτι της 97 αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Questo bisogna Ok. C'era un errore Α, είχα ένα λάθος εγώ στον δικό στη λίστα ψηφοφορίας. Λοιπόν, ψηφίζουμε το δεύτερο τμήμα της 97. Publishing από το 2008. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα λοιπόν της 97 αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίες, απορρίπτεται. 98. Αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίες, Απορρίπτεται. 99 και 100 μπορούμε να τα ψηφίσουμε μαζί. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνονται. 101. Αρχίζει η ψηφοφορία. 100, ε, πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 102. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 103 χωριστή ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα. Αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 104. Αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 105. Αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 106. Αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 108 αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. 109 αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. 112 αρχίζει η ψηφοφορία. 100... Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. 113. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία του εισηγητή αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Προφορική της κυρίας Γκρέσλε αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. 115 και 116 θα ψηφίζουμε μαζί, αρχίζει η ψηφοφορία. Όχι. Α, μία πρόταση ήταν, δεν θέλετε. Καλά. 115 λοιπόν ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Εκατόν δεκαέξι ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. 117. Ψηφίζουμε. Πέρασε ψηφοφορία εγκρίνεται 119 ψηφίζουμε πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται 120 αρχίζει ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται 121 αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. 123 αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. 124 αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 125 αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 126 αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 127 αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 128 αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 129 αρχίζει η ψηφοφορία Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. Οι 130 με 133 αν ψηφίσουμε unblock, αν συμφωνείτε. Ψηφίζουμε λοιπόν. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 134 αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. 135 αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. 139. 139 ψηφίζουμε. Πέρα στις ψηφοφορίες εγκρίνεται. 140 και 141 τις ψηφίζουμε μαζί. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρα στις ψηφοφορίες εγκρίνεται. 142 αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. αν θέλετε τις 143, 144 και 145 τις ψηφίζουμε μαζί. Όχι, όχι. Ε. Λοιπόν, 143 ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 144 ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας, εγκρίνεται. 145 αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας, εγκρίνεται. 149 αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας, εγκρίνεται. 150. Ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Προφορική τροπολογία του κυρίου Ήταλα. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 146 αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. Η κυρία Χέρτζοκ. Ζητώ συγγνώμη να υπενθυμίσω στους συναδέλφους σοσιαλιστές στην 1647 ε, και 48 υπάρχει ένα λάθος. Οπότε είμαστε κατά. Ζητώ συγγνώμη που παίρνω τώρα το λόγο. Ούτω ή άλλω δύο ψηφοφορίε θα γίνουν. Συμφωνούμε με το περιεχόμενο, δεν συμφωνούμε με τον τόπο όπου θα μπουν. 147 λοιπόν αρχίζει ψηφοφορία. Πέρες ψηφοφορίες. Απορρίπτεται. 148 αρχίζει ψηφοφορία. Πέρες ψηφοφορία εγκρίνεται. 152 αρχίζει η ψηφοφορία. Α, αποσύρθηκε, αποσύρθηκε αυτή, δεν την ψηφίζουμε. 153 αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 154 αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται. 155 αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 156 αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 157 αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Σχετικά με το σχέδιο της παραγράφου 106, ο κύριος Στάις έχει το λόγο. Συνάδελφοι, είχαμε ένα σχέδιο συμβιβασμού για την παράγραφο 106 μετά από διαβουλεύσεις χτες. Σας αποστήλαμε και ένα νέο κείμενο το εξής, αν εγκριθεί. Παράγραφος 106, το διαβάζω στα αγγλικά. Υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με το άρθρο 223 για τους κανονισμού, για τους ε, κανόνες αυτούς, κάθε ομάδα θα πρέπει να έχει σύστημα εσωτερικού ελέγχου. Όσο εκεί δηλαδή, το υπόλοιπο τμήμα όχι. Το υπόλοιπο τμήμα που διαβάζεται στον κατάλογο από το Introduce λοιπόν θα αντικατασταθεί με το Maintain και μετά το Control System θα διαγραφούν όλα τα υπόλοιπα στοιχεία. Ωραία. Ψηφίζουμε όλα όσα είπε ο κύριος Στάες. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Για τον συμβιβασμό 2, α, μπορούμε να ψηφίσουμε χωρίς να τα πει ο κύριος Τάις. Λοιπόν, ψηφίζουμε τον συμβιβασμό 2. Πέρα στις ψηφοφορίες, απορρίπτεται. Εκατόν αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίες, εγκρίνεται. 160 αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 161 και 162 τα ψηφίσουμε μαζί. Αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνονται. 163 αρχίζει ψηφοφορία. Πέρα στις ψηφοφορίες. Απορρίπτεται. 164. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορίες. Απορρίπτεται. 165. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 166. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. 167 αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. 168 αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. 169 αρχίζει η ψηφοφορία. 100 πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται 170 αρχίζει η ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται Unblock 171-173 αρχίζει η ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας απορρίπτονται 174 αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 175 αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 176 αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται 177. Όχι, αποσύρθηκε. 178. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 179. Αρχίζει. Πέρας. Εγκρίνεται. Εκατόν Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 181 αρχίζει η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. 182. Αρχίζει η ψηφοφορία, πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Αρχίζει 183. 183 έλεγα. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. Ο κύριος Τάς για τις παραγράφους 135, 135α και 135β. Συνάδελφοι, υπήρχε μια μεγάλη σειρά τροπολογιών που αναφέρονταν στις μεταφορές στα αυτοκίνητα, στα οχήματα και από πλευρά των φιλελευθέρων σε ό,τι αφορά και τα ποδήλατα από το ΕΛΚ για την ε, υποστήριξη της, και ε, την ενίσχυση της ε, των ε, αστικών επικοινωνιών και προσπάθησα με την τροπολογία τη συμβαστική τρία να αναφέρω όλες αυτές τις διαδάξεις. Ελπίζω να σας βρει σύμφωνος αυτή η πρόταση. Eh, Ψηφίζουμε. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα 135 και 135α. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρα τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. εγκρίνεται. τριάντα β χωρίς την παρένθεση που έχουμε στο τέλος. Αρχίζει η ψηφοφορία. εγκρίνεται. Για την παρένθεση τώρα. Πέρα τις ψηφοφορίες. Απορρίπτεται. Η ε, κυρία Γκρέσλε, ναι, έχουμε μία μικρή παρανόηση ψηφίσαμε την 135 Β. Είναι λίγο δύσκολο να τα κρατήσουμε τη σειρά στο σημείο αυτό, στο κατάλογο ψηφοφορίας. Ποιο ψηφίσαμε, το Α ή το Β. Ή θα ψηφίσουμε τώρα το Α ή το Β. Εμείς για το πρώτο τμήμα ψηφίσαμε το 135 και το 135α. Μετά ε, ψηφίσαμε το 135β χωρίς την παρένθεση και μετά ψηφίσαμε τη φράση που είναι μέσα σε παρένθεση και η οποία δεν πέρασε. Ωραία, καταλάβατε. Προχωράμε. Ok. Emendamento 190. 190. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 191 αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. Μαζί 192-193 ψηφίζουμε. Όχι. Ωραία. Ε, τώρα ψηφίζουμε 192 αρχής ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίες. Απορρίπτεται. 193 αρχής ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίες. Εγκρίνεται. 194 αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 195. Αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 196. Αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία με χωριστά τμήματα 197 αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίες, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα της 197 αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίες, εγκρίνεται. 198 ψηφίζουμε πέρα στις ψηφοφορίες απορρίπτεται 199 αρχίζει ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίες απορρίπτεται 200 αρχίζει ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίες Απορρίπτεται. 201 αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. 202 αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε συνολικά το ψήφισμα. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίες. Εγκρίνεται. 17 υπέρ 4 κατά και Ευχαριστούμε τον κύριο Στάις. Θέλετε να πείτε κάτι κύριε Στάις. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε που με επενείτε για τη δουλειά που έκανα. Μπορώ να διαπιστώσω ότι το μωρό μου δεν έχει γεννηθεί καν. Πρόκειται για ένα μωρό το οποίο στην αρχή το είχαμε ρίξει και τώρα πάμε σε ένα κείμενο στην Ολομέλεια με το οποίο ως εισηγητής Είμαι πολύ σίγουρος, εξ ονόματος και της ομάδας μου, σχηματίστηκε και μέτωπο από ό,τι είδα και από τις μικρές ομάδες ε, στο Κοινοβούλιο. Θα προσπαθήσω να υποβάλω και συμβολικές ε, ε, τροπολογίες εξ ονόματος των μικρών ομάδων για να υποδείξουμε και την κριτική στάση που τηρούμε έναντι του προπολογισμού. Ευχαριστούμε τον κύριο Στάες, ο κύριος η κυρία Γκρέσ. Ευχαριστώ, αγαπητέ Μπάρτ. Φυσικά τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Από το 2007 έχει αλλάξει όλος ο κόσμος σε ό,τι αφορά τον προϋπολογισμό και καλό θα ήταν αυτό να αποτυπώνεται ε, στην έκθεση. Πολλά από αυτά που έχεις ε, σχολιάσει δεν ισχύουν πλέον. Γι' αυτό θα ήθελα να είχαμε αφιερώσει λιγότερο χώρο και χρόνο σε ό,τι αφορά το θεωρητικό υπόβαθρο και τη θεωρητική κριτική, να είχαμε επικεντρωθεί πιο πολύ σε συγκεκριμένα στοιχεία περιεχομένου, γιατί υπάρχουν σε αυτό το κοινοβούλιο πάρα πολλά συστήματα, στοιχεία κριτικής. Θα ήθελα να τα έχουμε αναφέρει όλα αυτά. Ήμουν μόνη μου. Έχουμε συμφωνήσει πλέον από, επί αλλά λυπάμαι που δίδεται η εντύπωση ότι δεν ισχύουν αυτά που γίνονται στο κοινοβούλιο, στο Δεν μπορώ να επιτρέψω λοιπόν αυτή την εντύπωση να συνεχίσει να υπάρχει. Θα ήθελα πραγματικά επικοδομητικά να προσπαθήσουμε στο κοινοβούλιο να ρυθμίζουμε ό,τι πρέπει να ρυθμίζεται. Ο κύριος ε, Χατζημαρκάκης. καταρχά αγαπητοί, είναι συγχαρητήρια για το καινούργιο κούρεμα. Πολύ ωραίο. Και σου πάει. Δεν μιλάμε για θεωρητικό υπόβαθρο και υπερβολική ανάπτυξη του ε, θεωρητικού υπόβαθρου. Μιλάμε για κάποια πράγματα τα οποία πραγματικά έχουν κάποια σχέση και τα στηρίζουν και οι μικρές ε, ομάδες και γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι είναι καλό το γεγονός ότι ο εισηγητής είπε ότι κάποια στοιχεία θα προσπαθήσει παρόλα αυτά να τα περάσει και στην Ολομέλεια, να τα συζητήσει και με τις μεγάλες ε, ομάδες, για να μην είμαστε μικροί κατά των μεγάλων και εν ώψη των νέων εξελίξεων να αποτυπωθούν όλα αυτά στην ε, έκθεση και πραγματικά ευχαριστώ ε, τον εισηγητή γι' αυτό. Mm, Σας ευχαριστώ κύριε Τσορνέσκι. Είναι γεγονό ότι το ψήφισμα μετά τις τροπολογίες έχει τη μορφή που έχει. Ακούσαμε τα σχόλια και του εισηγητή και των άλλων συναδέλφων. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να αρνηθούμε ότι πρόκειται για μια διαφορετική έκθεση σε σχέση με τις προηγούμενες εκδόσεις. Μου φαίνεται ότι ο έλεγχος του προπολογισμού στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει βελτιωθεί. Είναι σαφώς καλύτερος από ότι ήταν στην κατάσταση, η κατάσταση πριν από πέντε χρόνια, στην αρχή της προηγούμενης θητείας. Δεν μπόρεσα να υποστηρίξω όμως την έκθεση στην παρούσα μορφή. Κυρία Χέρτσοκ, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρο, Ευχαριστώ και τον ε, κύριο Στάς, ο οποίος έθιξε πολλά θέματα και πολλά θέματα καταφέραμε να τα επιλύσουμε. Αλλά θα συμφωνήσω με όσους είπαν ότι τα τελευταία χρόνια έχει βελτιωθεί η διαδικασία ελέγχου του προϋπολογισμού και το βασικότερο μήνυμα είναι ότι εντός ε, της διαδικασίας ε, ιστορικού ελέγχου θα πρέπει να σημειώσουμε βελτιώσεις προβάλλατε και υποβάλλατε πολλές προτάσεις, κύριε Στάς, τις οποίες απορρίψαμε, αλλά και εκεί σημειώσαμε πρόοδο, γιατί μας έδωσε αυτή την ευκαιρία να, σκεφτούμε τι θα κάνουμε στο μέλλον και πώς μπορούμε να λάβουμε στο μέλλον αποφάσεις. Έχουμε μια διαδικασία η οποία έχει τεθεί πλέον σε ε, εξέλιξη και η οποία θα πάρει το δρόμο του. Κύριε Στάς, σας συγχαίρω, κάνετε μεγάλη πρόοδο και νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια θα μπορέσουμε, τα επόμενα χρόνια θα μπορέσουμε να επιλύσουμε τα ανοιχτά αυτά θέματα που παραμένουν. Νομίζω ότι πετύχαμε ό,τι μπορούσαμε να πετύχουμε. Σε ό,τι αφορά τις τροπολογίες τώρα για την Ολομέλεια, θα έλεγα να υπάρχει περαιτέρω εξέλιξεις. Chairman. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι το ερώτημα που ανακύπτει εδώ είναι κατά πόσο μας ικανοποιεί αυτή η εξέλιξη Είμαστε βέβαιοι ότι οι δαπάνες, τα κονδύλια του Ευρωπαίου Φορολογούμενου δαπανώνται σωστά. Αυτό θα πρέπει να μας απασχολεί. Συμφωνώ λοιπόν με την έκθεση του κ. Στάς. Αποδεικνύει ότι πολλά ακόμα πρέπει να πετύχουμε πέρα από αυτά που έχουμε ήδη πετύχει. Καλή πρόοδο, καλή εξέλιξη, αλλά δεν μα αρκεί αυτό που έχουμε πετύχει. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σόντεγκάρτ. Ευχαριστώ. Πλέον η έκθεση είναι διαφορετική. Σε 36 τομείς έχουν αλλάξει λιγότερο ή περισσότερο σημαντικά πράγματα. Η έκθεση αυτή λοιπόν έχει αλλάξει τελείως σε σχέση με την αρχική έκθεση. Σας ευχαριστώ όμως για την έκκληση αυτή που μας απευθύνατε για την περαιτέρω υποβολή ε, τροπολογιών στην Ολομέλεια. Λοιπόν, δεν υπάρχουν άλλες τοποθετήσεις. Προχωράμε με την απαλλαγή 2008 απόδοση χρηματοπιστωτική διαχείριση και έλεγχος των οργανισμών. Πριν προχωρήσουμε, το λόγο έχει η κυρία Ματιού. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εμείς ε, Προχωράμε στην ψηφοφορία της απαλλαγής για τους οργανισμούς και ζητώ να την υπερψηφίσουμε. Θέλουμε όμως να υπάρξει μία βελτίωση στη διαχείριση. Υπ' αυτήν την έννοια λοιπόν η έκθεση πρωτοβουλίας έχει ορισμένα χνάρια γενικών ε, προσανατολισμών. Παρακαλώ λοιπόν για, τη 2000, για το 2008 να αναβάλουμε την ε, απαλλαγή της ΕΠΟΛ. Παρ' όλα αυτά ε, έχουμε ελπίδες ότι θα επανορθώσουμε την κατάσταση χάρη στο σχέδιο δράσης ε, που θα εκτελέσει ο Διευθυντής του Οργανισμού και το Διοικητικό Σύμβουλο του Οργανισμού. Το βλέπετε το σχέδιο στο παράρτημα της έκθεσης. Ε, θα δούμε εν ώψη της επόμενης ψηφοφορίας ποια θα είναι τα αποτελέσματα του σχεδίου δράσης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τον επικοδομητικό διάλογο που είχαμε και ευχαριστώ και την γραμματεία όλος ιδιαιτέρως ε, για την αφοσίωση που έδειξε στις εργασίες της. Ευχαριστώ και προτείνω να αρχίσει ψηφοφορία. Ευχαριστώ κυρία Ματιέ. Προχωρούμε στην ψηφοφορία. για το ψήφισμα. Είστε έτοιμοι? Ψηφίζουμε λοιπόν το έγγραφο ENE. E. Είναι το ΙΤΕ με νέα. Είστε έτοιμοι? Τροπολογία 1. Αρχίζει η ψηφοφορία. Αρχίζουμε. Είστε έτοιμοι. Ξαναρχίζουμε. Λοιπόν, τροπολογία 1. Αρχίζει η ψηφοφορία. τη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 2. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τρία. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τέσσερα. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Πέντε. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Έξι. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Εφτά. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίες. Απορρίπτεται. 8. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 9. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 10. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτω. 11 αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψυχοφορίες. Εγκρίνεται. 12 αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψυχοφορίες. Εγκρίνεται. 13 προφορική τροπολογία. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 14. Αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίες. Απορρίπτεται. Έχουμε μία προφορική τροπολογία του κυρίου Σταυρακάκη. Έχετε το λόγο αν θέλετε. Θέλω να υποβάλω μία προφορική τροπολογία Συγκεκριμένα θα ήθελα να προσθεθεί στο τέλος του κειμένου της ε, παραγράφου 15α της, ε, της κυρίας Κρέσλερ το ε, απόλυτο κείμενο, το διαβάζω στα αγγλικά. But notes also that the agencies receive payments after the authorized work has been concluded and paid for, rapporteurs, etc., and therefore some cash holdings are essential in each case. Ευχαριστώ πολύ. Possiamo andare avanti? Possiamo votare? Να ψηφίσουμε. Ωραία, το ψηφίζουμε όπως τροποποιήθηκε. Λοιπόν, αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 16. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. 17. Αρχής ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. 18. Αρχής ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. Και εδώ έχουμε μία προφορική τροπολογία του κυρίου Σταυρακάκη πάντα Έχετε το λόγο κύριε Σταυρακάκη. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να υποβάλω μια προφορική τροπολογία στην τροπολογία της κυρίας Κρέσλερ με αριθμό 19 και στο τέλος του κειμένου προτείνω να προσθεθεί το ακόλουθ, η ακόλουθη παράγραφος. Διαβάζω στα αγγλικά. Notes, however, that the number of the decentralized agencies increased from 11 in 2000 to 29 in 2010, which is corresponding to 0.102% of the total EU budget in 2000 and 0.477% in 2010. Ευχαριστώ πολύ. Ψηφίζουμε τη 19. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 20. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 21. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Ψηφίζουμε μαζί την 22 και 23. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρα της ψηφοφορίες. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε τώρα το, το τροποποιημένο ψήφισμα. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 19 υπέρ, 4 κατά 2 αποχές. Ευχαριστούμε κυρία Ματιού. Πάμε τώρα. Έχουμε όλα τα, τους, όλους τους υπόλοιπους οργανισμούς και δίνω το λόγο στην κυρία Ματιού. Eh, Θέλετε να μιλήσετε ή να ψηφίσουμε. Προτείνω να ψηφίσουμε, Πρόεδρε, γιατί άμα στα, σταθούμε σε κάθε οργανισμό, ούτε το απόγευμα, ούτε το βράδυ θα τελειώσουμε. Ψηφίζουμε λοιπόν το item 10. Για το τσεντεφόπ ψηφίζουμε. Αρχίζει η ψηφοφορία για την απαλλαγή. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Για το κλείσιμο των λογαριασμών αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ψήφισμα. Λοιπόν, unblock τις 2, 7, 6 και 5 ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνονται. Τελική ψηφοφορία του ψηφίσματος αρχίζει. Πέρας. Εγκρίνεται. 19 υπέρ 2 κατά. το CDT. Απαλλαγή. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρες ψηφοφορίες. Εγκρίνεται. για το κλείσιμο των λογαριασμών. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 3, τροπολογία 1. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρασε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τελικό ψήφισμα. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 21 υπέρ, 2 κατά, μία εποχή. Πάμε στην Ευρωπαϊκή Ακαδημία Αστυνομίας. Σε πόλ. Αρχίζει η ψηφοφορία για την απαλλαγή. Πέρασα. Εγκρίνεται. για το κλείσιμο των λογαριασμών. Πέρασε. Μπορούμε να ψηφίσουμε τη γνωμοδότηση 3, 4, 5 όλα, όλες μαζί. Λοιπόν ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. Ένα. Τροπολογία 1. Αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τελικό ψήφισμα. Αρχής ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με 24 υπέρ, έναν κατά. Λοιπόν, οργανισμός ελέγχου της Αγίας σε, σε, σε α, αρχής ψηφοφορία για την απαλλαγή πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. Για τους λογαριασμούς αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. Τελικό ψήφισμα υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Λοιπόν, Passiamo adesso Europea per la Ψηφίζουμε τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ανοικοδόμης, τον ΕΡ. Απαλλαγή. Αρχής ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Λογαριασμοί, Αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τελικό ψήφισμα, τροπολογία 1, αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 2. Αρχίζει. Πέρας ψηφοφορίας, εγκρίνεται. Τελικό ψήφισμα. Αρχίζει ψηφοφορία, πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Πάμε στην ΕΑΣΑ για την αεροπορική ασφάλεια. Συνολικά η απαλλαγή. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συνολικά λοιπόν για το κλείσιμο των λογαριασμών. Πέρας ψηφοφορίας. Για το τελικό ψήφισμα, εάν συμφωνείτε, να τα ψηφίσουμε όλα μαζί τα... Δηλαδή, Ψηφίζουμε. 1, 2, 3, 7 και 4. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 1 αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τα σημεία 5 και 6 μαζί. Αρχίζει ψηφοφορία. Πέρες Εγκρίνεται. Τελικό ψήφισμα. Αρχίζει ψηφοφορία. Αρχής ψηφοφοριες Εγκρίνεται. 20, 21, 1 και μία αποχή. Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Πρόληψη και τον Έλεγχο των Ασθενειών, το SDC. Αρχίζουμε με την απαλλαγή. Πέρας ψηφοφορίες. Εγκρίνεται. Λογαριασμοί. Αρχίζει. Πέρας ψηφοφορίες. Εγκρίνεται. Τα πρώτα τρία θα ψηφίζουμε μαζί ένα πέντε έξι. Α, συγγνώμη. Γνωμοδότηση 1. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. Πέντε αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Έξι αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ένα αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 3, 7 και 4 μπλοκ, αν δεν έχετε αντιρρήσεις. Λοιπόν, ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συνολική ψηφοφορία, λοιπόν. Votazione chiusa. Approvato. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. 23 υπέρ ένας κατά μία αποχή. Πάμε στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τις Χημικές Ουσίες ε, για την απαλλαγή. Άρχεται η ψηφοφορία παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται 21 ψήφοι υπέρ, ε, μια ε, αποχή, δύο κατά. Τώρα για το κλείσιμο των λογαριασμών, άρχεται η ψηφοφορία παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται. Το νούμερο 2 τώρα, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Το 5, υπέρ. Ε, συγγνώμη, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Το 1, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 1. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Το 3. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία για το ψήφισμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας εγκρίνεται 23 υπέρ 2 κατά και μία αποχή. Τώρα περνάμε στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος. Η απόφαση για την απαλλαγή. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται 24 υπέρ 1 κατά μία αποχή. Για το κλείσιμο των λογαριασμών άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στο 1 και 4 μαζί. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνονται. Τώρα 2 και 3 ομαδών. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτονται. Τελική ψηφοφορία για το ψήφισμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται 24 υπέρ, 1 κατά μία αποχή. Τώρα, Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων, ε, απόφαση για την απαλλαγή, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται 23 υπέρ 2 κατά μία αποχή. Πρόταση για το κλείσιμο των λογαριασμών. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τώρα, ομαδών να πάρουμε τα πρώτα τρία. Τρία, ένα και δύο. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνονται. Τροπολογία 1. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Αρχή. Πέρας. Εγκρίνεται. 4. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Το 5. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται 22 υπέρ 2 κατά μία αποχή. Τώρα, Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τα Ναρκωτικά και τις Τοξικομανίες, ε, απόφαση για την απαλλαγή, έρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται 23 υπέρ 1 κατά μία αποχή. Για το κλείσιμο των λογαριασμών τώρα, έρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. τις δύο πρώτες γνωμοδοτήσεις. Ένα και τρία μαζί παρακαλώ. Άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνονται. Τροπολογία 1. Άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνονται. Συνολική ψηφοφορία για το ψήφισμα. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. 22 υπέρ, μία ψήφος κατά, μία αποχή εγκρίνεται. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων. Απόφαση για την απαλλαγή. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται 21 ψήφοι υπέρ, μία κατά, μία αποχή. Τώρα κλείσιμο λογαριασμών. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνονται. Τώρα, γνωμοδότηση υπαρθμών 1. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Γνωμοδοτήσεις 2 και 5 μαζί. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνονται. Τροπολογία 1. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται. Γνωμοδότηση 6. Ψηφίστε. Πέρας. Εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται 23 ψήφοι υπέρ, μία κατά. Ευρωπαϊκός Οργανισμός ε, για τη Θαλάσσια Ασφάλεια, ΕΜΣΑ. Άρχεται ψηφοφορία για την απαλλαγή. Πέρας. 24 ψήφοι υπέρ, μία κατά. Για το κλείσιμο των λογαριασμών τώρα, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τώρα, ομαδών, γνωμοδοτήσεις 6, 1 και 2. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνονται. Τροπολογία 1. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία. Παρακαλώ. Ψηφίστε. Πέρας. 24 ψήφοι υπέρ, μία κατά εγκρίνεται. Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια των Δικτύων Πληροφοριών. για την Ασφάλεια. Ε, απόφαση για την απαλλαγή άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται 20 ψήφοι υπέρ, μία κατά, δύο αποχές. Για το κλείσιμο των λογαριασμών τώρα, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Ε, τροπολογία υπαριθμών 1. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία. Παρακαλώ ψηφίστε. Πέρας. Εγκρίνεται. 23 ψήφοι υπέρ, 2 κατά, μία αποχή. Ευρωπαϊκός ε, Οργανισμός για τους Σιδηροδρόμους. Η απόφαση για την απαλλαγή. Παρακαλώ ψηφίστε. Πέρας εγκρίνεται 21 ψήφοι υπέρ, μία κατά, μία αποχή. Ε, τώρα για το κλείσιμο των λογαριασμών, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Ε, γνωμοδοτήσεις όλες μαζί, 1, 2 και 5. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνονται. Για το ψήφισμα, τελική ψηφοφορία παρακαλώ. Πέρας. 20 ψήφοι υπέρ, μία κατά εγκρίνεται. Ε, Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για την Κατάρτιση, απόφαση για την απαλλαγή, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 19 υπέρ μία κατά μία αποχή εγκρίνεται. Για το κλείσιμο των λογαριασμών τώρα, ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται. Γνωμοδοτήσεις 2 και 3 μαζί. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνονται. Ε, ψηφίζουμε τώρα για το ψήφισμα, παρακαλώ. Πέρας. Ε, εγκρίνεται 20 υπέρ 2 κατά μία αποχή. Ευρωπαϊκός Οργανισμός ε, για την Ασφάλεια και την Υγεία στο χώρο εργασίας. Απόφαση για την απαλλαγή. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται 20 υπέρ, 1 κατά, μία αποχή. Για το κλείσιμο των λογαριασμών τώρα. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται για τη γνωμοδότηση 2 και 3 μαζί. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνονται. Ε, τροπολογία 1. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Ψηφίστε. Πέρας. Εγκρίνεται. Γνωμοδοτήσεις 4 και 5 μαζί. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνονται. Τελική ψηφοφορία, παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται 20 υπέρ 2 κατά μία αποχή. Τώρα Πάμε ε, στον οργανισμό ανεφοδιασμού Ευρατόμ. Ε, η πρόταση για την απαλλαγή. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται 19 ψήφοι υπέρ μία αποχή για το κλείσιμο των λογαριασμών. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται 20 ψήφοι υπέρ, 2 κατά. Τώρα, Eurofound, Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Όρων Διαβίωσης και Εργασίας. Απόφαση απαλλαγής. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται 21 ψήφοι υπέρ 2 κατά μία εποχή. Ε, πρόταση για το κλείσιμο των λογαριασμών. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 1 υπέρ. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ε, θα ψηφίσουμε μαζί τις νομοδοτήσεις 2, 3 και 6. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνονται. Άρχεται η τελική ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνονται 21 ψήφοι υπέρ κατά μία αποχή. Eurojust. Ε, η απόφαση για την απαλλαγή. Ε, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας εγκρίνεται 21 ψηφί υπέρ μία κατά μία αποχή. Τώρα για το κλείσιμο των λογαριασμών άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Ε, εγκρίνεται. Ε, ε τώρα γνωμοδοτήσεις 1 και 3. Μαζί ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνονται. Τροπολογία 1. Ε, ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε συνολικά για το σχέδιο. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 21 ψήφοι υπέρ μία κατά μία αποχή. Τώρα, ε, οργανισμός για τα θεμελιώδη δικαιώματα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως για την απαλλαγή συνολικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας εγκρίνεται 21 ψήφοι υπέρ μια κατά. Ε, για το κλείσιμο των λογαριασμών. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Ε, ψηφίζουμε μαζί τις νομοδοτήσεις 1 και 3. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνονται. Άρχεται η τελική ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται 20 ψήφοι υπέρ, 2 κατά και 1 αποχή. Τώρα, Ευρωπαϊκό Οργανισμό ε, για την Διαχείριση τη Επιχειρησιακή Συνεργασία στα Σύνορα των Κρατών Μέλων τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω, Frontex. Ψηφίζουμε για την απαλλαγή. Παρακαλώ. Πέρας εγκρίνεται 19 ψήφοι υπέρ 2 κατά μία αποχή. Ε, τώρα για το κλείσιμο των λογαριασμών άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Ε, γνωμοδότηση 1 υπέρ. Ε, συγγνώμη, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 1 τώρα, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Γνωμοδοτήσεις 5 και 6 μαζί. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνονται. Άρχεται η τελική ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται 20 ψήφοι υπέρ 2 κατά μία αποχή. Ε, τώρα, Ευρωπαϊκή Αρχή Εποπτείας. GSA. Ε, πρόταση για την απαλλαγή. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται 20 ψήφοι υπέρ μία κατά μία αποχή. Ε, για το κλείσιμο των λογαριασμών άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Ε, τροπολογία 1 τώρα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Ε, ψηφίζουμε για την έκθεση συνολικά, παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται. 20 ψήφοι υπέρ 2 κατά μία αποχή. Ευρωπαϊκή Κοινή Επιχείρηση, ΤΕΡ, για την ενέργεια σχάσης. Ε, ψηφίζουμε πρώτα για την απαλλαγή. Άρχεται η ψηφοφορία ε, πέρας. Εγκρίνεται 18 ψήφοι υπέρ 2 κατά μία απόχη. Ε, τώρα για το κλείσιμο των λογαριασμών άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Ε, τροπολογία 1. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Άρχεται η τελική ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται 20 ψήφοι υπέρ, 2 κατά μία εποχή. Κοινή επιχείρηση Σέζαρ. Ε, ψηφίζουμε για την απαλλαγή πρώτα, παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται 19 υπέρ 1 κατά 2 αποχές. Ε, τώρα για το κλείσιμο των λογαριασμών. Άρχιτε ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Ε, ψηφίζουμε τους νομοδοτήσεις 1, 2, 3, 5, 7 ομαδών. Παρακαλώ, άρχιτε ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνονται. Τροπολογία 1. Άρχιτε ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Ε, τροπολογία 2. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Γνωμοδοτήση 6. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε για την έκθεση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 20 ψήφοι υπέρ μία κατά δύο αποχές. Ευχαριστούμε την κυρία Ματιέ για τις εργασίες της. Τελειώσαμε και νωρίτερα. Μπορούμε να πιούμε και καφέ. Τα λέμε το απόγευμα και πάλι. Γεια σας.